Good afternoon everybody and thank you very much for coming to the GUE NGL press briefing. Um... Καλώς ήρθατε στην συνέντευξη τύπου της GUE. Να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμερ, πρόεδρο της ομάδας. Ja, um, guten Tag, Damen und Herren. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα ε, υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα και όταν υπάρχουν και προκύπτουν εξελίξεις, αυτές προκύπτουν ραγδαία. Ανακοινώσαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα στην εδρίαση της ομάδας μας ότι σήμερα θα λάβουμε ένα έγγραφο που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευόμασταν με βάση αυτό, με βάση την επόμενη Κυριακή όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση των διαφόρων θεσμών. Και σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί υποτίθεται θα είχαμε το χρόνο να τοποθετηθούμε επ' αυτού του εγγράφου. Τώρα όμως προέκυψε μία ανακοίνωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή δημοσιεύτηκε ε, στα μέσα ενημέρωσης. Ε, είναι ένα εκτεταμένο σχέδιο. Στο τέλος αυτού ακολουθεί και μία δήλωση στον τύπο και από εκεί μπορούμε να συνάγουμε το τι θα προκύψει. Βεβαίως πρέπει να σας πω εμείς δεν είχαμε καμία δυνατότητα να τοποθετηθούμε επ' αυτού του εγγράφου και είναι και πολύ δύσκολο ε, να τοποθετηθεί κανείς πάνω σε αυτό εκ των υστέρων εφόσον αυτό το κείμενο προκύπτει από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποια σχόλια γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σοβαρά πρέπει να δούμε λιγάκι τη διατύπωση να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά Καταλήγω λοιπόν στο εξής. Ο κύριος Τούσκ προτείνει να ικανοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ προχωρημένο βαθμό, τα αιτήματα του κυρίου Κάμερον. Άρα δηλαδή ο κύριος Τούσκ δίνει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθοριστικά θέματα όλη τη την ύπαρξη και το θέμα της ενοποίησης όλα αυτά τα αποσύρει σε μεγάλο βαθμό και κατά την άποψή μας αυτό το γεγονός θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη συμβίωση των Ευρωπαίων πολιτών. Και μας, ε, μας ενδιαφέρει η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, και κατά το παρελθόν επικρίναμε ότι η Μεγάλη Βρετανία επέλαξε το opting out σε πολλά θέματα είτε σε ειδικέ ε, λύσεις ε, για τις εκπτώσεις ε, και σε πολλά άλλα θέματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε γιατί σε τελική ανάλυση είναι ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας και στο πλαίσιο αυτής, γιατί θα πρέπει να ικανοποιήσουμε τόσο πολύ τα αιτήματα του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κινδυνεύει η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση που προκύπτει ότι σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να προκύψει ένας μηχανισμός ο οποίος ε, θα μπορούσε να ισχύει όχι μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και για άλλες χώρες. Ε, Παραδείγματο χάρη είναι Παραδείγματο χάρη λοιπόν οποτεδήποτε θα προκύπτει μεγάλη ροή μεταναστών από άλλα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση αυτή ε, θα μπορούσε το θυγόμενο κράτος να καταφύγει στο παράγωγο δίκαιο και στο πλαίσιο και ακριβώς λόγω παραγώγου δικαίου θα έχει το δικαίωμα να ε, αναστέλει κοινωνικές παροχές μέχρι και τέσσερα χρόνια αυτό ελέγχθη. Εμείς όμως διαφωνούμε με αυτό και θέλω να ελπίζω ότι και άλλα κράτη-μέλη θα δηλώσουν τη διαφωνία τους. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ακριβώς αυτός ο περιορισμός, ε, παραδείγματος χάρη του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης, ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών, δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι αν υπάρξει περιορισμός ε, σε αυτό το δικαίωμα ότι θα γίνει δεκτό από κάποια κράτη-μέλη. Για να υπάρξει μια τέτοια αλλαγή, δηλαδή να εισαχθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, απαιτείται ομοφωνία. Και ελπίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν κράτη που θα πούνε όχι δεν συμφωνούμε. Γιατί αν υπάρξει κάτι τέτοιο κατ' ουσίαν θα σημαίνει αναστολή της κοινωνικής Ευρώπης, καταγγελία της αρχής ε, ότι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από ποια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται απολάβουν των ιδίων δικαιωμάτων όπως και όλοι οι άλλοι δηλαδή ε, ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αρχή της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης αν λοιπόν ισχύσουν όλα αυτά ε, θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και σε τελική ανάλυση όσον αφορά αυτή την πρόταση αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ε, οικονομικό χώρο όπου ισχύουν διαφορετικά νομίσματα και κράτη τα οποία δεν είναι στην Ευρωζώνη, θα πρέπει και αυτά να μπορούν να αποφασίζουν εξίσου για σημαντικά θέματα. Έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προβεί ε, σε τέτοιου είδους αλλαγές και πρέπει να σας πω ότι αμφιβάλλω κατά πόσον αυτά που είπε ο κύριος Τούσκ τα εννοούσε σοβαρά. Αύριο λοιπόν θα ακούσουμε την ε, άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο πλαίσιο της συζήτησης για την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής θα ακούσουμε πώς αιτιολογούν αυτές τους τις ε, απόψεις και επίσης ε, θα ακούσουμε και πώς θα συσταθεί η απαραίτητη νομική βάση. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχει μια σειρά ανοιχτών θεμάτων αλλά όπως σας είπα αυτά που ακούτε σήμερα είναι η πρώτη μας αντίδραση σε αυτά που μας ε, σερβίρισαν ε, την τελευταία μισή ώρα. Και εμείς θα τοποθετηθούμε από αυτόν ως πολιτική ομάδα σήμερα και αύριο θα εκδώσουμε μια επίσημη τοποθέτηση η οποία τοποθέτηση θα τεθεί από τους ε, διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου, τους περίφημους Sherpers και κατόπιν τούτου να περιμένετε ότι ως πολιτική ομάδα θα επικρίνουμε την διαδικασία η οποία δεν μας επιτρέπει σε μας και σε άλλες ε, μικρότερες ε, πολιτικές ε, ομάδες δεν μας επιτρέπει να επηρεάσουμε τη διατύπωση αυτού του εγγράφου. Η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής. Σε πρώτη φάση έχουμε τρεις εντεταλμένους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι ε, διαπραγματευτές αν θέλετε οι ε, Γκαλτιέρη, Μπροκ και Φεχόφστατ, ε, αυτοί θα αναλάβουν να προβούν στην απαραίτητη αξιολόγηση και μετά θα πάρουμε τη δική τους πρόταση αυτών των τριών ανθρώπων και εκεί πια δεν ξέρουμε πώς θα παρισφρήσει η δική μας θέση. Εμείς πώς θα επηρεάσουμε ε, την απόφαση που θα έχουν παρουσιάσει αυτοί οι τρεις κύριοι. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το πούμε αυτό στον πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά ε, θα καταθέσουμε τις ε, απόψεις μας. Αυτά είχα καταρχήν να σας πω. Αυτή είναι η πρώτη μας αντίδραση. Όσον αφορά στις ε, προτάσεις που κατατέθηκαν, αυτά είχαμε να σας πούμε ε, και κατά την άποψή μου όλα αυτά δείχνουν ότι αποστασιοποιούμεθα από καθοριστικές θεμελιώδεις αρχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πράττει ε, ο επικεφαλής μιας πολύ σημαντικής, ενός πολύ σημαντικού θεσμού της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το παρελθόν ας μην ξεχνάμε ότι οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές, στην εξασφάλιση της εργασίας, οι περιορισμοί των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων, περιορισμός της ε, συλλογικής αυτονομίας, όλα αυτά ε, οδηγούσαν στο να προκύπτουν συγκεκριμένες περικοπές σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Τι θέλουμε να πούμε, θέλουμε να πούμε ότι οι μετανάστες που έρχονται και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί θα υποστούν περικοπές και αυτομάτως θα προκύψει αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και των γηγενών, των υπηκόων μιας ε, χώρας. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου ε, θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς ε, την αντίδραση των Βρετανικών Συνδικάτων και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ε, θα ζήσουμε μια πολύ ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση. Αυτά είχα να σας πω εγώ και ευχαριστώ πολύ. Στέλιο παρακαλώ. Εγώ θα σας πω δύο λόγια για την ε, ΤΙΖΑ, ε, την Διεθνή Συμφωνία για τις Υπηρεσίες, όπου θα συζητηθεί αύριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εγκρίνει ε, ή θα απορρίψει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία διαπραγματεύεται εκ μέρους των 28 κρατών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης την, ε, τη συμφωνία αυτή. Εμείς είμαστε αντίθετοι με τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι η ήδη υπάρχουσα συμφωνία είναι, η, η GATS είναι αρκετή. Αν χρειαζόταν εξυγχρονισμό θα μπορούσαμε να την εξυγχρονίσουμε. Ε, είναι μια συμφωνία την οποία τη μόνη που θέλουν και την προωθούν είναι οι μεγάλες πολυεθνικές ε, εταιρείε. Είναι φανερό ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τη θέλουν. Ε, γι' αυτό και η κυρία Ρέντινγκ στην, στην προσπάθειά της να, που είναι η συγγήτρια, στην προσπάθειά της να πετύχει ε, την ε, κάποια συνένεση ε, έκανε μια σειρά από θετικές παραχωρήσεις για τις οποίες όμως αμφισβητούμε πάρα πολύ ότι θα, την, θα τις πάρει υπόψη της η, η Κομισιόν. Ενώ υπόθηκαν και υπόθηκαν τρομερά πράγματα στη διάρκεια της ε, συζήτησης στο Ευρω... χτες στη διάρκεια της συζήτησης και ενώ ε, Ρέντιν είχε πει διάφορα πράγματα τι απάντησε η κυρία Μάρστρομ στο τέλος τι είπε θα σας το διαβάσω Thank you for the ε, report No problem at all for the Commission We will Για την Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται τη συμφωνία ΤΙΖΑ ε, με τον ίδιο τρόπο λες και εμείς είχαμε συμφωνήσει. Δεν ε, σκέφτονται καθόλου να αλλάξουν ε, ε, τη συμφωνία αυτή και ούτε να πάρουν υπόψη τους και αυτές τις μικρές διαφοροποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. έχουμε προτείνει μια σειρά από ε, τροποποιήσεις στο, στο, τροπολογίες στο σχέδιο που έχουμε προτείνει αλλά περισσότερα ε, στο σχέδιο που προτείνεται. Ε, έχουμε κάνει τροπολογίες, αλλά περισσότερο για αυτές θα σας πούμε στις 4 η ώρα που έχουμε εδώ μια συνέντευξη τύπου ειδικά ε, για την ΤΙΖΕ και μπορούμε να σας πούμε αναλυτικά και το παρασκήνιο και για τις... εδώ δεν είναι και για το παρασκήνιο και για, το, και για τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Ευχαριστώ. Thanks, Ευχαριστούμε, Στέλιο. Ο Φάμπιο Ντεμάζη για τον εταιρικό φόρο και την δέσμη μέτρων. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται σε συνέντευξεις τύπου, δηλαδή θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, δημοκρατικό υποψήφιο, τον αντίπαλο ε, της ε, Χίλερ Κρίντον για τις για την υποψηφιότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, στη θέση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτείων. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι οι εργαζόμενοι φέρνουν σε μεγάλο βαθμό το φορολογικό βάρος ενώ πολυεθνικές όπως η Google δεν καταβάλουν καθόλου φόρους και έτσι λοιπόν αυτό αποδεικνύει ότι με φορολογικές υποσχέσεις δεν μπορεί κανείς ε, να κερδίζει εκλογές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στι ΗΠΑ ε, και στην Ευρώπη που είναι εξοργισμένοι για το ότι οι πολυεθνικές ε, ξεφεύγουν, ξεγλιστρούν. Φαίνεται όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξάγει τα σωστά συμπεράσματα. Γιατί τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο πακέτο, στην τρίτη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με βάση τις προτάσεις τα σκάνδαλα όπως το LuxLeaks ε, δεν μπορούν να αποφευθούν με αυτή τη δέσμη μέτρων που έχει κατατεθεί. Και θέλω να καταστήσω σαφές το εξή. Υπάρχει καταρχήν ο φραγμός στους τόκους. Φραγμός στους τόκους. Δηλαδή το κατά πόσον μία χώρα μπορεί κέρδη από τόκους να τα εμβάσει σε χώρα με χαμηλή φορολογία. Αυτό γίνεται κατά 30% και αυτό είναι το ανώτατο όριο αυτού που έχει επιτρέψει ο ΩΣΑ. Δηλαδή, αν πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν ισχυρίζεται ότι έχει καθοριστική θέση στην αντιμετώπιση της ε, διαφθορά και του αθέμητου ανταγωνισμού λέει ψέματα γιατί έπιασε μόνο το ελάχιστο από αυτά που υποσχέθηκε όσα. Δεύτερον, ως αριστερή εμεί ε, στο Κοινοβούλιο θέλουμε να τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα. Ε, το κατά πόσο μπορεί μια ε, εταιρεία να μεταφέρει τα κέρδη σε όχι. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει το, ο φόρος να είναι ενιαίος, να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο παντού, ενοποιημένο τρόπο η εταιρεία, το unitary taxation. Δυστυχώς όμως αυτή τη μέτρων η ε, Κομισιόν το εγκατέλειψε. Ξέρετε γιατί, γιατί επιτρέπεται η θηγατρική μιας ε, πολυεθνικής ε, να μεταφέρει τα κέρδη της σε φορολογικό παράδοσο και εκεί να φορολογείται μόνο το 60% του προσποριζόμενου κέρδους. Και η Ιρλανδία, ας πούμε, που έχει συντελεστεί 12,5% υποτίθεται είναι απόλυτα εντάξει η πολυεθνική να μεταφέρει τα κέρδη της σε αυτήν την χώρα. Υπότιτλοι υπάρχουν ε, πολλοί που πληρώνουν φόρους. Φαντάζομαι και εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ κανείς στην αίθουσα που να πληρώνει 5%, συντελεστή 5%. Ε, το βρίσκω απαράδεικτο οι γραμματείς να φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή από την Google. Ε, εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά περί θηγατρικών εταιριών, περί κερδών, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Εμείς ε, τα σώμεθα υπέρ της δημοσιοποίησης των ισολογισμών και των κερδών και η αποκάλυψη του Reuters ε, για τους ε, Βρετανούς ε, τραπεζίτες που δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου πόρους. Αν αυτό είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα δεν θα μπορούσε να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο και να πω και κάτι άλλο. Πριν από λίγο καιρό καταθέσαμε αγωγή στην Επιτροπή Τάξε η οποία ε, Επιτροπή έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και μπορείτε να τη βρείτε τις δηλώσεις της ε, και στη δική μου στον Λέμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμφωνία TTIP ε, ήταν πάρα πολύ περιοριστική και μόνο αυτό αλλά έσβησε και κάποιες πληροφορίες. Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά αυτή την αγωγή θα κερδίσουμε στο δικαστήριο και στις 26 Απριλίου όταν ο whistleblower the tour θα δικαστεί στο Λουξεμβούργο. Εγώ προσωπικά θα πάω στο Λουξεμβούργο και θα είμαι εκεί παρόν γιατί θέλω να εκπέμψω το μήνυμα από τη δική μου την πολιτική ομάδα ότι δεν είναι δυνατόν να κάθονται ε, στο εδόλιο οι κατηγορούμενοι, οι whistleblower και ο κύριος Γιούνκερ ε, χαρούμενος και αφελής και ανέμελος να περιδιαβαίνει εδώ στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου και να πίνει καφέ. Ευχαριστούμε. Θα εμπειρωτήσεις. Από το Reporter μια ερώτηση για την κυρία Τσίμερ. Εάν κατάλαβα καλά, δεν θεωρείτε την διαδικασία για την βρετανική διευθέτηση που επίκειται δημοκρατική. Εσείς τι διευθέτηση προτείνετε, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συζητηθεί και πώς θα θεωρούσατε τη διαδικασία δημοκρατική. Ποια είναι η συγκεκριμένη πρότασή σας. Ich kann das ganz kurz sagen. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ε, το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει τώρα. Μας είπαν ε, ότι ξέρετε πρόκειται μόνο για τεχνικές ε, ψηφοφορίες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο θα είναι αναγκασμένο να δεχθεί ό,τι αποφασιστεί στις 17 και 18 του μήνα. Και επειδή προφανώς δεν προβλέπονται αλλαγές στις συνθήκες, αλλά μέσα από το δευτερογενές δίκαιο θα καταβληθούν προσπάθειες να περάσουν ρυθμίσεις όπου θα αναφέρεται ότι με τις ε, συνακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις ε, αυτές οι ρυθμίσεις θα συμπεριληφθούν στο δευτερογενές δίκαιο ε, με αυτόν τον τρόπο θα τελείσουν να ρυθμίσουν τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό όμω είναι πολύ αμφίβαλο αν θα επιτευχθεί ως στόχος η Βρετανική κυβέρνηση ο κύριος ε, Κάμερον αναφέρει ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα εθνικά κράτη θα πρέπει να είναι μικρότερος. Και εδώ βλέπω την εξής προσέγγιση, ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ολοκλήρωση και εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δική μας θέση. Κατά την άποψή μου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπό τους ε, αρχηγούς ε, κυβερνήσεων στο Συμβούλιο να επικρατήσει η συμφωνία και να παραγωνίσουν ε, το κοινοβούλιο. Κάπου θα επιτευχθεί ένα συμβασμός και μετά θα μας πούνε αυτό είναι δεχτείτε το και τέλος. Yes. Ευχαριστούμε άλλες ερωτήσεις αν και δεν είναι το θέμα σας, ε, θα σας παρακαλούσα για ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση του περιορισμού κοινωνικών επιδομάτων στην περίπτωση της Βρετανίας. Διότι, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι σοβαρό το θέμα. Η Βρετανία είναι ίσως ο πρώτος και σίγουρα ένας από τους πρώτους προορισμούς για νέους Έλληνες που ε, αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βλέπετε εκεί κάποιο πρόβλημα ή κάποιον κίνδυνο. Ε, κατά τη γνώμη μου ο κίνδυνος δεν αφορά ε, μόνο ή κυρίως ε, τους Έλληνες ε, υποψήφιους μετανάστες αφορά άλλους μετανάστες από άλλες χώρες, φτωχότερες της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τους πρόσφυγες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο παραβιάζει τους βασικούς κανόνες της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των πολιτών στις, στις ευκαιρίες. Δημιουργούνται πολίτες δύο κατηγοριών. Οι πολίτες οι Βρετανοί και κάποιοι άλλοι και οι, οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας είτε ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η μέλη η Βουλγαρία ή η Ρουμανία ή και η Ελλάδα και σε, στους Βρετανούς. Αυτό είναι τελείως έξω από τις αρχές, δεν υπάρχει. Άρα αν δεχτούμε αυτές τις παραχωρήσεις, την πραγματικότητα ε, αυτό αποτελεί τη χαριστική βολή στις ευρωπαϊκές ε, αξίες. Και αργά ή γρήγορα θα έχει επιπτώσεις και στην ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κλείνουμε εδώ τη συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευση. Η συντονίστρια ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Και να επενθυμίσουμε τη συνέντευξη τύπου στην ίδια αίθουσα στις 4 η ώρα το απόγευμα, ειδικά για την Τίζα. Και όχι με εκπροσώπους μόνο της Γκουελέου κ. Κούλογλου, αλλά και με άλλους συναδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες.